Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε καθυστερήσει. Καθυστερούμε μάλλον την αρχή. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κατάλογο ψηφοφορίας των φιλελευθέρων, ο οποίος δεν έχει έρθει εγκαίρως. Και γι' αυτό ζητώ από όλους τους συναδέλφους να κάνουν λίγη υπομονή. Για να μπορέσουν και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοι να ψηφίσουν κανονικά. Λοιπόν, μόλις τώρα μου ήρθε το έγγραφο με τον κατάλογο των φιλελευθέρων. Ελέγξτε αν δουλεύει η κάρτα σας, βάλτε την κάρτα σας στη σεισμή για να δούμε αν πράγματι είναι, ε, ανάβει το φωτάκι και δουλεύει γενικά το σύστημα. Bene, ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες για τη σύσταση προς το Συμβούλιο για την 65η Συνέλευση του Ηνωμένων Εθνών. Παράγραφος 1, σημείο α, έχω την τροπολογία 17 Μελανσόν. Ποιοι είναι υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ.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 Κατά. Δεκτή. Η 30 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 20, 32 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη 42 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 46. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 46. Αρχίζουμε. «58 ψήφισαν, Δύο δεν ψηφίζουν, 31 υπέρ, 29 κατά δεκτή. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην προφορική τροπολογία υπαρίθμ 1, την οποία ψηφίζουμε κατά διαίρεση, πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικός έλεγχος να γίνει για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας προφορικής 1. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουν 62. Κάποιος έχει χτίσει το λόγο. Now it's on. Okay, thank you. Mr. Um, Άναψε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το να ψηφίσουμε το τμήμα 2 χωρίς να έχουμε ψηφίσει το τμήμα 1 δεν στέκει. Παρακαλώ να ελέγξετε αν ε, η ψηφοφορία επί του τμήματος 1 ήταν όντως αρνητική, γιατί εγώ είχα αντίθετη εντύπωση, οπότε ή στην προφορική τροπολογία 1, χρειαζόμαστε όλο το κείμενο για να έχει νόημα η ψηφοφορία επί του δεύτερου μέρους που είναι χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι συνάδελφοί μας της ΓΚΟΕ. Οπότε μπορούμε να ελέγξουμε το πρώτο μέρος και μετά να ψηφίσουμε επί του δεύτερου. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Θέλετε να υπάρξει λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος και για τα δύο καμάτια και όχι μόνο για το πρώτο. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα της προφορικής 1. Ξεκινάει η ψηφοφορία. ...64 ψηφίζουν, αλλά 61 μόνο ψήφισαν. 35 υπέρ, 29 κατά, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα τώρα, της προφορικής 1. Ξεκινάμε. 31 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Θα ψηφίσουμε τώρα τη συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ της 6ης. Κατά. Δεκτή. Συνεχίζουμε με τη συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. οι ενδιάμεσε καταπίπτουν. Την 57. Ποιοι είναι υπέρ 57. Κατά. Απορρίπτεται. Ή μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 57. Αρχίζουμε. 34 υπέρ 27 κατά δεκτή. Η 58 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ της 58. είναι κατά. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 60 υπέρ. Κατά. Δεκτή νομίζω. 61 υπέρ κατά απορρίπτεται. 62 είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Προφορική υπαρίθμου 2 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 8 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. 65 υπέρ κατά δεκτή 66 υπέρ κατά δεκτή συμβιβαστική 9 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 67 ποιοι είναι υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 67. Ξεκινάμε. «33 υπέρ 30 κατάθεκτη. 69. Όχι, η 69 έχει καταπέσει γιατί ψηφίσαμε τη συμβιβαστική 9. 70, ποιοι είναι υπέρ της 70, κατά. Απορρίπτεται. 71, υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 10, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 77, ποιοι είναι υπέρ. Συγγνώμη. 76, ποιοι είναι υπέρ Κατά. Απερίφθη 76. 77 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 78. Ψηφίζουμε. Τέλος. 29 κατά 34 υπέρ. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν σας βλέπω καλά και μετά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικούς ελέγχους και καθυστερούμε. 79 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 80 λοιπόν. Ψηφίζουμε. Για την 80. Ψηφίσαν 62. 41 κατά. 21 υπέρ. Απορρίπτεται. 81. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά απορρίπτεται 84 υπέρ κατά απορρίπτεται 85 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά απορρίπτεται και σκέψη έχουμε τη 2 ποιοι είναι υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. 35 κατά, 27 υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, δεκτή. Στην 4 θα υπάρξει καταδιέρεση ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ της κατά, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα, αποσύρθηκε το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, δεκτό. Η 5. Ποιοι είναι υπέρ της 5. Κατά. Δεκτή. Προφορική υπαρίθμη 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα. Στην 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 13. Ψηφίζουμε. «32 υπέρ, 31 κατά». Γίνεται δεκτή με μία ψήφο διαφορά. 14 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. 15 κατά. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε τέσσερις τροπολογίες από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Καταρχάς την πρώτη της ανάπτυξης ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Η β μικρό ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Γ μικρό ποιοι είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη γάμα μικρό της ανάπτυξης. Ξεκινάμε. Κάποιος δεν ψηφίζει γρήγορα. Λοιπόν. 31 κατά, 34 υπέρ. Δεκτή. Και την δέλτα μικρό της Επιτροπής Ανάπτυξης ψηφίζουμε. Κατά. Δεκτή. Τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Ξεκινάμε. Ένας δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Υπάρχει κάποιος που έχει βάλει την κάρτα του αλλά δεν ψηφίζει. Λοιπόν, 59 κατά, 4 αποχές, κανείς, ε, συγγνώμη, 59 υπέρ, δεκτή λοιπόν. Συγχαρητήρια στον Λαμπστόφ. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία τώρα. Θέλετε το λόγο κύριε Λάμστορφ. Ευχαριστώ. Σύντομα να ενημερώσω του συναδέλφους πρώτα απ' όλα πως η συνεργασία με την Επιτροπή ανάπτυξη, ήταν εξαιρετική, αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Θα πάω τώρα στο Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για μια σύσταση προς το Συμβούλιο και φέτος για δεύτερη φορά έχουμε μια πρόσκληση να παρουσιάσουμε αυτές τις ε, προτεραιότητες. Έχουμε λοιπόν ένα διάλογο μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις στρατηγικές προτεραιότητες για τον ΟΗΕ. Είναι μια θετική εξέλιξη που ήθελα να αναφέρω. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάνθρο. Και πάμε τώρα στην ψηφοφορία για τι ειδικέ πτυχέ τη προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχουμε την ε, παράγραφο 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αγκρίνεται. Τροπολογία 2 στην παράγραφο 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβασμός 1, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, πάμε στο συμβασμό 3, υπέρ, κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5. Συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 9, όχι, γιατί το 3 ενεκρίθη. 10, υπέρ, κατά, Δεν ήταν σηκώνω τα χέρια, οπότε άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 10. Άρχεται. 65 δελτία, 61 ψήφισαν. Λείπουν λοιπόν, 4. Τρεις. Λείπουν... Όχι, λείπουν τρία. Τρεις. Σας παρακαλώ τρεις καφέδες για τους συναδέλφους που δεν ψήφισαν. Να ξυπνήσουν. Σοφορία. Έληξε. 33 υπέρ, 27 κατά εγκρίθηκε. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 11 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά απορρίπτεται. 14. Α, στη 12 θέλετε έλεγχο. Στη 12. Ωραία, 12. Άρχεται η ψηφοφορία. ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 12. Άρχεται. 65 δελτία, 63 ψήφισαν, 64 ψήφισαν. 1, 2, 3, λίγη ψηφορία. 29 κατά 33 υπέρ εγκρίθηκε. Τροπολογία 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 16 σε δύο τμήματα. Όχι, ο συμβασμό 1. Πάμε στην 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 συμβατή με την 19 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 21 καταπίπτει. Πάμε στην 22. Α, καταπίπτει. Πάμε στην 23. Υπέρ. 23 ψηφίσμα Υπέρ. Κατά. πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 23. Αρχή. Πάντα λείπει ένας. 30 κατά 32 υπέρ. Περνάει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της έκθεσης άρχεται. 65 δελτία, 62 ψήφισαν. Έληξε. 57 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία που αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχέση με την Γενική Αμερική. Εισηγητής ο κύριος Αλαφράνκα. Ξεκινάμε με την τροπολογία Μελανσόν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 32, που είναι ταυτόσημη 33, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 34, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 Α, θέλετε στην 36 άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 36. 63 τις κάρτες δεν ψήφισαν 30 κατά 30 υπέρ απορρίπτεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 119 Μελανσόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41. Ταυτόσημη 42. Όχι. Ε, Γλωσσική φύσεως δεν ε, ψηφίζουμε. Συμβασμός 8. Υπέρ. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Κύριε Νανούλητσα, θέλετε το λόγο. Ναι, ε, ήθελα να, κάνουμε και άλλη μία ψηφοφορία συμπεριλαμβάνοντας τη βία λόγω φύλου μια συμβαστική πρόταση ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Μέγερ που δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμβασμό. Άρα θέλω να ψηφίσουμε ε, επιπλέον αυτό το σημείο. Να ακούσω και την άποψη του εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι αυτό που προτείνει η κυρία Λούνατσεκ είναι προφορική τροπολογία. Το θέμα δηλαδή της βίας λόγω φύλου καλύπτεται απόλυτα στις ιδεολογικές σκέψεις. Κατ' του κανονισμού, επειδή πρόκειται για προφορική τροπολογία, δεν νομίζω ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Θα, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όπως προβλέπεται μέσα στον κατάλογο ψηφοφορία. Βεβαίω, ε, είναι σωστή η παρατήρησή σα, αλλά θα πρέπει να, να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Συμφωνείτε με τον κύριο Σαλαφράγκα και όχι με την, πρόταση την προφορική πρόταση τροπολογία, ε, για να δω τι γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμό, σα υπενθυμίζω, αρκεί ένα άτομο. Α, μάλιστα, ωραία, εντάξει. Αρκεί λοιπόν που διαφωνείτε εσεί, μάλιστα. Δεν μελέτησα το, τον κανονισμό για τι επιτροπέ, ήξερα μόνο ότι γίνεται στην Ολομέλεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Συμβασμό 8. Υπέρ. Κατά. Από... Εγκρίνεται. 46 γλωσσική φύση. 120. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 47 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβασμό 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στο 49 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβασμό 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 51 υπέρ κατά εγκρίνεται 52 υπέρ κατά εγκρίνεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβασμός 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 58 υπέρ απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εγκρίνεται Περνάμε στο 61 υπέρ κατά δεκτή 62 όχι καλύπτεται η 62 65 υπέρ κατά απορρίπτεται 63. Ποιοι είναι υπέρ της 63. Κατά. Απορρίπτεται. 64. Ή θέλετε ηλεκτρονικός έλεγχος να γίνει για την 63 λοιπόν. Κλείνει η ψηφοφορία. 33 κατά, 28 υπέρ. Απορρίπτεται. 64. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά απορρίπτεται 68 υπέρ κατά νομίζω απορρίπτεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά δεκτή 73 προφορική τροπολογία 73 υπέρ έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Λούνατσεκ. Αυτό το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι η 70 θα πρέπει να ψηφιστεί. Ο κύριε Σαλαφάνκα. Αυτή τη στιγμή γίνεται δεκτή συμβιβαστική τροπολογία, σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει είναι και αντίθετη με την προφορική τροπολογία. Καλά. Συνεπώς η 70 καταπίπτει και περνάμε στην 73 χωρίς προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την 73 σκέτη λοιπόν, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 75 και 122 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Προφορική 4 υπέρ. Κύριε Σαλαφάνκα. Όχι, δεν, ε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν συμφωνούμε. Allora, si Είστε κατά λοιπόν τη ψηφοφορία αυτής. για, να μας εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να ε, γίνει δεκτή μια προφορική τροπολογία που ήδη βρίσκεται στον κατάλογο της προφορίας που δεν είναι έτσι ε, μια τροπολογία που εμφανίστηκε ε, τώρα. Ναι, πρώτα απ' όλα γιατί το θέμα των, ε, των περιφερειακών ζωνών είναι εκτός θέματος συγκεκριμένη περίπτωση. Καλώς δεν ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική 4 και ψηφίζουμε την 123. Α, κάποιος άλλος έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι ομάδες θα αποφασίσουν ε, κατά πόσον ε, θα ψηφίσουμε ή όχι. Δεν μπορεί ο εισηγητής ε, μια τροπολογία που ήδη έχει γίνει δεκτή από τη γραμματεία της Επιτροπής δεν μπορεί να πει δεν την ψηφίζουμε. Διαβάζω λίγο αυτά τα οποία λέγει ο κανονισμός που διέπει την ψηφοφορία. Οι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί προφορικά στι επιτροπέ μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία εκτό και αν μέλο τη επιτροπή είναι αντίθετο. Είναι ένα μέλο αντίθετο, συνεπώ δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Λυπάμαι για αυτού που διαφωνούν, αλλά το κείμενο νομίζω είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται άλλη ερμηνεία. Λοιπόν, 123 λοιπόν, θα ψηφίσουμε την 123, ξεκινάμε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 76 του εισηγητή υπέρ, κατά, δεκτή. 124 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, δεκτή. 78 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 79 υπέρ. Α, όχι, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 78. Λοιπόν, μέχρι την 62, 62 μάλλον είναι εδώ, που θα ψηφίσουν 35 υπέρ, 27 κατά δεκτή. Περνάμε τώρα στην 79. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 80 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 82 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, δεκτό. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 83. Αν θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για το τρίτο τμήμα της 82, ψηφίζουμε. sono sempre due che non votano. 60 eh, chiudiamola. 37 <laughs> 37 κατά 26 υπέρ απορρίπτεται. 83 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά δεκτή. Φτάνουμε τώρα στην 87 του εισηγητή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 87 υπέρ κατά δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεκτή. 88 υπέρ κατά δεκτή. 89 υπέρ κατά δεκτή. 90 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 91 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Φτάνουμε στην 17 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 94 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά δεκτή. 98 τώρα. Υπέρ. Κατά δεκτή. 99 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 127 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 100 και 101 υπέρ. Ακαλύπτονται. Μάλλον από τη συμβιβαστική 18. Έκανα λάθος. Δεν θα ψηφίσουμε την 100 και 101. Καλύπτονται από τη 18. Φτάνουμε στην 128 υπέρ κατά, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, δεκτή. 102 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, Δεκτή. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 129 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά δεκτή. 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. 113 γλωσσική. Οι 5 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 6 θα την ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 6 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 8 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Σε δύο τμήματα τώρα, σε τρία τμήματα μάλλον, θα ψηφίσουμε την 12 υπέρ του πρώτου τμήματος της 12. Κατά. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 14. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα γίνεται μια διευκρίνηση. Θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία 6 και αν απορριφθεί θα ψηφίσουμε το 15. Κύριε Σαραφάνκα. Διαφωνούμε την προφορική τροπολογία, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον κανονισμό ψηφίζουμε την τροπολογία 15. Υπέρ. Όσοι, έχει υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, απορρίπτεται λέω. Έχω την εντύπωση. Για σηκώστε και λίγο τα χέρια, γιατί η γυμναστική δεν κάνει κακό. 16 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά. 115 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται 18 υπέρ κατά. Απορρίπτεται 19 υπέρ κατά. Απορρίπτεται 20 υπέρ κατά. Εγκρίνεται 21 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 4. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26. Όχι, όχι. Καλύπτει από την 6. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη 28. Έχουμε την προφορική τροπολογία 7. Ψηφίζουμε μαζί με την τροπολογία 28. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 29. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία προφορική 8. Υπέρ, κατά, να κάνουμε έναν έλεγχο. Κύριε Σαραφράκα, θέλετε το λόγο. Όχι. Θα έκανα λοιπόν ένα έλεγχο στην προφορική τροπολογία 8, γιατί δεν είδα τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφορία. 65 δελτία, 63 ψήφισαν. Κλείνει η ψηφορία. Στην προφορική τροπολογία αυτή, 63 ε, ψήφισαν, 26 υπέρ, 37 κατά. Τροπολογία 1 ε, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Αλλά έπρεπε να το μαντέψω, έτσι. 9 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε Ε, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Αλλά πριν ο κύριος Σαλαφράγκα ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Σαλαφράγκα. Eh, κύριε Πρόεδρε, πήραμε πολύ καθυστερημένα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Έφτασε χτες το βράδυ αργά. Ειλικρινά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των σημείων που μας υποβάλλει η Επιτροπή Ανάπτυξης ήδη καλύπτει από την έκθεση. Προτείνω μόνο μία ή δύο δεν συμπεριλαμβάνονται προτείνω στα μέλη της Επιτροπής για να είμαστε συνεπείς να απορρίψουμε όλα τα σημεία της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ, λέει η κυρία Λούνατσεκ, με τον εισηγητή. Λυπάμαι. Στην Επιτροπή Ανάπτυξη χθε ε, έγινε συνεδρία και ψηφοφορία. Μπορεί να, ε, να έπρεπε να, έχουμε, να έχει οργανωθεί καλύτερα ο χρόνο ψηφοφορία. Αλλά βεβαίω ε, λογικό είναι να, πάει, να φτάσει το βράδυ. Γι' αυτό λέω να, ψηφίσουμε μία προς μία, μία, προς μία τις ε, τροπολογίες. Πολλά από αυτά τα σημεία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του εισηγητή. Λυπάμαι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, Πρόεδρε κύριος Μέγερ και μετά Βίγκενιν. Και εγώ δεν συμφωνώ, διότι πράγματι πρέπει να ψηφίσουμε ε, όλες αυτές τις τροπολογίες, μία-μία της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης. Είναι αλήθεια ότι έφτασαν αργά, αλλά να, να θυμίσω στον εισηγητή ότι και χτες στην αρχή της συνεδρίας πήραμε τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τα οργανωτικά προβλήματα, αλλά τι να γίνει έτσι έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε. Βίγκενιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρα από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω πως πρέπει να σεβαστούμε τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης. Οπότε εμείς θα θέλαμε να γίνει η ψηφοφορία όπως ε, είναι εδώ πέρα. Ωραία. Τότε θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες μία-μία. Ξεκινάμε με την παράγραφο 1. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ε, ε, ε, εντάξει, συμβολικό είναι ο έλεγχο. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Αλλά βλέπετε, είχαν σηκωθεί τα χέρια. Μία θα κάνουμε, έτσι, ένα έλεγχο. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στην παράγραφο 1. 65, δελτία 64 ψήφισαν. Α, 32. Α, μα είχατε δίκιο, είχατε δίκιο, είχατε δίκιο. Α, ωραία. Απορρίπτεται, αλλά Τότε θα κάνουμε όλε τι ψηφοφορίε. Υποκλίνομαι. Τι να σα πω, λέει ο πρόεδρο. Μάλιστα, δικό μου λάθο. Σηκώστε τα χέρια. Παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Για μένα απορρίπτεται, αλλά ξέρω, θέλετε έλεγχο. Ε, το φανταζόμουν, το φανταζόμουν. Ηλεκτρονική ψηφορία στην παράγραφο 2. Ωραία, τι ωραία. Σήμερα παίζουμε με, τα... με την ηλεκτρονική ψηφορία, λέει ο πρόεδρος. Α, αυτή τη φορά δύο δεν ψηφίζουν. 66, 64. 31 απορρίπτονται, 28 υπέρ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Υπέρ, κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ο πρόεδρος... Τι το λέτε για πλάκα ή αλήθεια. Α, έλεγχος. Ωραία, εντάξει. Παράγραφος 3. Ωραία. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία σε όλες τις τροπολογίες, έτσι. Παράγραφος 3. Άρχεται ψηφοφορία. Παράγραφος 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάντα κάποιος δεν ψηφίζει. Έγλυξε. Α, πέρασε αυτή τη φορά με δύο. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, λέει ο πρόεδρος, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τρία ε, ε, επόμενη παράγραφος. 34 λέει πρόεδρο. Όχι, δω συγγνώμη, διορθώνει παράγραφο 4. Όχι, 34 ήταν η ψηφοφορία. Η ψήφη λέει ο πρόεδρο. 4 λοιπόν, ψηφίζουμε. «37 προς 27 απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, παράγραφος 5». Για ένα λεπτό, να, κλείσουμε αυτή τη ψηφοφορία και μετά θα σα το λόγο. Να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε τη ψηφοφορία. Ε, αν λείπει η ψηφοφορία σου, θα τη λάβουμε υπόψη ψήφο, θα τη λάβουμε υπόψη με, ε, ξεχωριστά. Μικρόφωνο. Υπάρχει το κουμπί που το πατάμε και μιλάμε. Στα δεξιά, στα δεξιά. Στο συγγνώμη πρόεδρε, επειδή εγώ είμαι ένα πληρωματικό μέλος, από ό,τι κατάλαβα το ΕΛΚΑ έχει... είναι πλήρε. αλλά θα ήθελα να μάθω, επειδή εδώ έχουμε ε, διαφορέ με μία-δύο ψήφου. Τι να κάνω, να ψηφίσω ή να μην ψηφίσω, έχω τη δυνατότητα. Αυτό θέλω να μάθω. Ωραία. Κοιτάξτε, ε, αυτός είναι έλεγχος των τεχνικών. Αν ο αριθμός των μελών ε, ε, του ΕΛΚ είναι, έχει καλυφθεί, δεν μπορείτε να ψηφίσετε γιατί θα θυμώσουν οι άλλοι. Α, κοιτάξτε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Μάλιστα. Παραβρέ, παραβρίσκεσαι, αλλά δεν μπορείς. Λοιπόν, 38, ε, ε, ε, πάμε στην 6 τώρα. Άρχεται ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία στην παράγραφο 6. Εντάξει, αν κάποιος κοιμηθεί, μπορείς. Απορρίπτεται, 53 με 12. Παράγραφος 7. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία στην παράγραφο 7. Λίγοι... 49 κατά 16 υπέρ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Άρχεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εδώ βλέπω υπέρ. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Έληξε. Α, 63 υπέρ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ομοφωνία. 9. Παράγραφος 9. Άρχεται στην παράγραφο 9. 55 κατά, 6 υπέρ, απορρίπτεται. Στη 10 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχη. «57 υπέρ 7 κατά εγκρίνεται». Ηλεκτρονική ψηφοφορία στην παράγραφο 11 αρχή Έληξε. 32 κατά 33 υπέρ εγκρίνεται. 12 υπέρ. Όχι, άρχεται, άρχεται. Να σας πρότεινα μπλοκ, αλλά ξέρω δεν θα συμφωνήσετε. 32 κατά 33 υπέρ. Εγκρίνεται. 13. Ηλεκτρονική ψηφορία αρχή. Πέρα 42 κατά 23 υπέρ. Απορρίπτεται. 14. Μα κάθε φορά ψηφίζεται διαφορετικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στη 14. Άρχεται. Έληξε. 48 κατά στα 16 υπέρ. Απορρίπτεται. 15. Παράγραφος 15. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ηλεκτρονική ψηφορία έληξε. 55 κατά 9 υπέρ απορρίπτεται. 16, παράγραφος 16, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχή. Πέρας. 32 κατά 31 υπέρ. Απορρίπτεται. 17, παράγραφος 17, αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην παράγραφο 17. 65, 33 ε, ε, υπέρ, 32 κατά, εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο τελικό ψήφισμα. Bene, 54. 54 υπέρ, μία ψήφος κατά, 9 αποχές. Συγχαρτήρια στον εισηγητή, συγχαρτήρια στη γραμματεία ε, που εργάστηκε πολύ σκληρά. Τελειώσαμε τις ψηφορίες, 5 λεπτά διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε 5 λεπτά. Περιμένουμε να ε, φύγουν από την αίθουσα οι συνάδελφοι που δεν ε, ενδιαφέρονται για το επόμενο θέμα.